Nous allons continuer notre euh, réunion après cette... Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, να συνεχίσουμε μάλλον κατά όπιν της κοινής συνεδρίασης που είχαμε με την Επιτροπή Αλλαγού του Προπολογισμού. Αν ε, συμφωνείτε, προτείνω μία μικρή τροποποίηση της ημερησίας ε, διάταξης ε, για να ε, έχουμε να δούμε την αντιλαγή αποψίων ε, με τον Πρωθυπουργό της Κεντρικής ε, Αφρικής στο τέλος του απογεύματος. Θα το δούμε ακριβώς πριν τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 5. Υπάρχουν σχόλια ή κάποιες αντιδράσεις. Αν όχι, εγκρίνεται η μερισσία οχι γκρινεται έτσι όπως τροποποιήθηκε. Και θα εγκρίνουμε τα πρακτικά για τη συνεδρία στις 18-19 Φεβρουαρίου και στις 18 19 Μαρτίου. Αν δεν υπάρχει κάποια διαφωνία κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Επίσης ε, θα εγκρίνουμε τις αποφάσεις και τις συστάσεις των συντονιστών της 19 της Μαρτίου. Έχετε όλοι στους φακέλους σας ε, τις συστάσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν ε, στις 19 Μαρτίου στη συνεδρίαση των συντονιστών. Αν έχετε σχόλια σχετικά με τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης θα πρέπει να τα γνωστοποιήσετε στη γραμματεία μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή συνεδρίαση. Αν όχι, θεωρείτε ότι εγκρίνονται. Δεν έχω συγκεκριμένες ανακοινώσεις ε, για σήμερα και θα ζητήσω την Επιτροπή αν θέλει να μας ανακοινώσει κάτι. Όχι. Από την πλευρά της Επιτροπής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση. Έχουμε μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφο Μπάστας. Θα βρείτε το σχετικό κείμενο στο φακελό σας. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Λουίς Βιέρα, συντονιστής της Task Force για την, ε, ε συντονιστής για τις επαφές με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω στο ερώτημα. Εγώ σήμερα το πρωί ήρθα από την νεαρινή συνάντηση της Παγκόσμιας Τράπεζας όπου ο πρόεδρος Κιμ έκανε μια παρουσίαση των σχεδίων του για το μέλλον αναφέρθηκαν βασικοί στόχοι που θα εγκριθούν τον Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα προσχέδιο στρατηγικής όπου η τράπεζα ε, επιβεβαιώνει τη βούλησή της να κάνει ορισμένα πράγματα για να μειώσει τη φτώχεια και να να... προωθήσει το sharing prosperity μια προσπάθεια δίκαιης κατανομής αν θέλετε ευημερία ή εν πάση περιπτώσει να βοηθηθεί τον, το 40% των πολιτών που βρίσκονται σε πολύ άσκημη κατάσταση. Είναι θέμα δικαιοσύνης και ισότητας Επίσης θα ήθελα να πω ότι μία από τις δεσμεύσεις του νέου Προέδρου της Τράπεζας είναι στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που πρέπει να γίνει να είναι να δουλέψει αν θέλετε σε, σε διάφορους τομείς της τράπεζας. Μοιάζει αυτό με το ερώτημά σας. Υπάρχει μια πολιτική... Ασφάλειας, διασφάλισης ε, γενική ή ειδική είναι μόνο για ορισμένες περιπτώσεις. Ε, για την τεχνική βοήθεια βεβαίως υπάρχουν ορισμένα μέτρα αλλά δεν ε, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο Program for Results και το Development Policy Lending εφαρμόζεται μοναχά στη τεχνική ποιες με στα πλαίσια ορισμένων ταμείων όπου α, παρέχεται ε, τεχνική βοήθεια. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι τα άλλα εργαλεία, τα καινούργια εργαλεία που δημιούργησε η τράπεζα δεν έχουν ασφάλεια, δεν έχουν κλίδες ασ, ασφάλειας. Η τράπεζα ξέρει πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο χρειάζονται και στη διαδικασία να αναθεώρησης των safeguards θα πρέπει να ε, ε, γίνουν οι συζητήσεις για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να εναρμονιστούν οι λεγόμενες δικλείδες ασφαλείας. Τώρα, Τώρα, κυρία Πρόεδρε, ίσως ε, εμείς μπορούμε να θέσουμε το ίδιο ερώτημα λέτε στην ερώτησή σας ε, ότι θα έπρεπε να θέσουμε το ίδιο ερώτημα στην, ε, στους διευθυντές των ε, ευρωπαϊκών προγραμμάτων θέσαμε το ερώτημα και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα θα γίνει μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών μεταξύ της ε, ε κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και των σχετικών στελεχών της τράπεζας και στις 15 Μαΐου έχουμε τους διευθυντές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία ούτω ώστε άμεσα να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να δείτε πώς βλέπουν την όλη διαδικασία αναθεώρησης των safeguards. Από άποψη χρόνο προγράμματος ε, πρέπει να πούμε ότι φτάνουμε στη δεύτερη φάση, είμαστε στη δεύτερη φάση της αναθεώρησης που Και θα ξεκινήσει από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο λοιπόν μια καινούργια σειρά διαβουλεύσεων οπότε και εκεί θα έχετε και εσείς και εμείς και όλοι τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις. Και για να τελειώνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ένα ρόλο μεσάζοντος αν θέλετε και συντονιστή αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά είμαστε μονάχα παρατηρητές ε, προνομιούχοι μπορεί ε, παρατηρητές αλλά κύριος ε, ο Επίτροπος ε, πηγαίνει στις συνεδριάζει στις τράπεζες αλλά δεν είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας δεν είναι μέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις αυτές Έχω μια ερώτηση συνέχιση. Θα ήθελα να ξέρω αν η Παγκοσμία Τράπεζα απαγορεύει τώρα τη χρηματοδότηση όλων των project, ε, ε, ξεκινώντας από την εκρίζωση, το land grabbing, δηλαδή όσοι στην Αιθιοπία ασχολούνται με τα βιοκαύσιμα και λειτουργούν κάτι τέτοιο ή στην Αιθιοπία ή σε κάποιε άλλε αφρικανικέ χώρε θα λάβουν βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα. Και δεύτερη ερώτηση, απαγορεύει η Παγκόσμια τράπεζα τη χρήση ε, των φορολογικών παραδείσων για την, ε, για την ίδια δραστηριότητα, τη δική της δραστηριότητα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αμέσω. Ε, η Παγκόσμια Τράπεζα προφανώς όπως εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα του grabbing, της εκρίζωσης είναι ένα σημαντικό θέμα για το μέλλον. στο πλαίσιο ενό ε, ανανεωμένου ενδιαφέροντος ε, για την συντηρητική ασφάλεια και την ανάπτυξη της υπαίθρου, την αγροτική ανάπτυξη. Φυσικά αυτό το land grabbing ε, θα μπορούσε πραγματικά να προκαλέσει μεγάλη συμφόρηση. Ε, πώς ξέρετε, εμείς υποστηρίζουμε τη ΦΑΟ και την Επιτροπή Επιστηστικής Ασφάλειας για όσα έχουν ήδη εκπονηθεί, για τις ε, κατευθυντήρες γραμμές που έχουν ήδη εκπονηθεί και για τη διάδοσή τους για το land grabbing. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω Θα έχετε βέβαια και την ευκαιρία να θέσετε αυτή την ερώτηση στους εκτελεστικούς διευθυντές, όμως ε, δεν πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση ναι ή όχι δηλαδή το land grabbing ε, πιθανότητα ή οι επενδύσεις, ε, ιδιωτικέ επενδύσεις ε, στη γεωργία. Για αυτά τα δύο είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μία σειρά μείγματος πολιτικών από θεσμική σκοπιά και σε ό,τι αφορά και την εμπλοκή των πληθυσμών, τη συμμετοχή των πληθυσμών. Επομένως είμαι σίγουρος ότι βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν συμφωνηθεί πρέπει να εργαστούμε επί της χάραξης μια πολιτικής αναπερίπτωση. Όμως επιμένω βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν συμφωνηθεί, των αρχών που έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να διασφαλίσουν αυτές οι αρχές αυτές ότι αυτές οι επενδύσεις ε, ωφελούν άμεσα τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα το σημείο 8 στην ημερησία διάταξη, την ανασυγκρότηση και τον αντιδημοκρατισμό του Μαλίου. Το Μαρτίο του 2012, πάνω από ένα χρόνο, είχαμε ένα πραξικόπημα στο Μαλί φέτος, στις 11 Ιανουαρίου 2013 ξεκίνησε μια νέα σύγκρουση στο μελί με την έναρξη της ε, γαλλικής στρατιωτικής επιχείρησης που επέτρεψε στο ε, στρατό, στο γαλλομαλικό στρατό να ξαναπάρει τον έλεγχο των ε, κύριων πόλεων της του βόρειου τμήματος της χώρας. Στις 29 Ιανουαρίου είχαμε την υιοθέτηση του χάρτη πορείας για τη μετάβαση που ε, υπογραμμίζει τις δύο κύριες αποστολές που έχει η κυβέρνηση μεταβατική να αποκαταστήσει την ακαιρεότητα την εδαφική και να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκες εκλογές. Ε, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ε, μεγάλες δυσκολίες ε, οργανωτικές και από άποψη ασφαλείας και επίσης Υπάρχουν δυσκολίες επειδή σιγά σιγά μειώνονται οι καλλικές δυνάμεις. Η κατάσταση παραμένει ζωτική σημασία σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Πάνω από 4.300.000 κάτοικοι του Μαλή χρειάστηκαν συγγνώμη, ανθρωπιστική βοήθεια το 2012, δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού από τον Απρίλιο του 2012 περίπου ε, μισό εκατομμύριο άνθρωποι ε, ε προσπάθησαν ε, να βρουν καταφύγιο στις γειτονικές χώρες ή στο ίδιο το μελή μεταξύ αυτών 65.000 ε, περίπου εκτοπίστηκαν ε, επίσης από τον Ιανουάριο φέτος. Η κατάσταση σε σχέση με το σοβασμό των ανθρωπίνων είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η κρίση έπληξε επίσης μέσω όλων χωρών την οικονομική παραγωγή και τις ε, βασικές δημοσίες υπηρεσίες. Μία πρόταση υπερφορικής ε, ερώτησης και μία πρόταση ψηφίσματος ε, θα υποβληθούν ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Σήμερα θα συζητήσουμε λοιπόν το ζήτημα αυτό και θα δώσω σε εσά το λόγο. Bon, alors, Monsieur Prada, D'accord, très bien. Donc, voilà, vous avez la parole pour Monsieur Préda. Voilà. Euh, oui, je prends la parole à la place. Μάλιστα, θα μιλήσω εκ μέρου του κύριου Πρέντα, γιατί μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Δεν μπορούσε να έρθει σήμερα το απόγευμα. Έτσι λοιπόν, θέλει να χαιρετήσει την ε, ε, εισαγωγή αυτού του θέματος ε, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου του Μαΐου για το θέμα της ανασυγκρότησης και του νομιμοκρατισμού του μελή καθώς το Μάιο θα λάβει χώρα μία συνάντηση δωρητών στις Βρυξέλλες. Επίσης χαιρετίζει τη γαλλική παρέμβαση για να υπερασπίσουν την εδαφική ακαιρεότητα και επίσης για την υπεράσπιση του ε, πληθυσμού θα ε, χρειαστούν συγκεκριμένες δράσεις από την πλευρά της Ένωσης, γιατί η ανοικοδόμηση του Μαλή σημαίνει ότι πρέπει να απαντήσουμε σε ε, προκλήσεις πολιτικές, ανθρωπιστικές που σχετιζόνται με την ανάπτυξη της χώρας. Ε, θα χρειαστεί καλύτερα στοχευμένη βοήθεια που να επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας και να υπάρχει καλύτερο συντονισμός με τους δωρητές. Η πολιτική διαδικασία επίσης είναι ζωτική για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τη χώρας χώρας. Ε, ε, πρέπει να υποστηριχθεί η οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας στη χώρα και να βρεθούν τρόπος να πιεστούν ε, οι αρχές έτσι ώστε να επιθεθεί μια σχετική ημερομηνία αναφοράς για τις εκλογές. Έχει γίνει διαπραγμάτευση και με την ΑΦΕΤ και για εξεσυμβαστικές τροπολογίες και για άλλες τροπολογίες και θα ήθελε ο κ. Πρέντα να καταλήξουμε σε ένα ισχυρό κείμενο που να καλύπτει συνολικά το πολύπλοκο ζήτημα του Μαλή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τα Ηνωμένα Έθνη μελετούν το ενδεχόμενο ψηφίσματος για την τοποθέτηση 12.600 ειρευτικών ε, δυνάμεων από την 1η Ιουλίου στην περιοχή ώστε να επιτραπεί στη Γαλλία να αποσύρει στα τα στρατεύματά τη. Εν τούτη, υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε όσον αφορά την δυνατότητα αυτών των δυναμεών την δυνατότητα μάλλον των Ηνωμένων Εθνών να εξεύρει τέτοιου είδου δυνάμει. Το ρήτημα είναι τι είδου ε, εκπαίδευση θα παράσχουν οι δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είδου συντονισμό προβλέπεται μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα είναι ο ρόλος της ε, ΣΕΝΤΑΟ Αφρικανικής Ένωσης από τον Ιούλιο και πέρα. αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, έχω και άλλες δύο. Ο κύριος Σαντόι. Thank Κυρία Πρόεδρε, είμαι επικεφαλή ε, του ΕΕΣ, του Τμήματος για την Δυτική Αφρική. Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι απλώς να παρασχεί ενισχύσεις. Θέλουμε να συμμετάσχουμε στην διαδικασία που καταστάσει τη κανονική ζωή στην περιοχή. Η δυνατότητα τη αφρίσμα είναι θέμα συζήτηση αυτήν τη στιγμή. Μελετούμε το θέμα αυτή τη στιγμή. Μια σχετική συνάντηση συντονισμού έγινε με τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και με την πολιτική διεύθυνση του ΟΗΕ υπό τον Έντμον Μιουλέ, βοηθό του Γενικού Γραμματέα, όπου συζητήσαμε ακριβώ τα συντονισμού συνειδητοποίησαμε και μάλιστα επιβεβαιώσαμε ότι έχουμε τις ίδιες ακριβώς ανησυχίες. Τώρα, οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής δράσης είναι ακριβώς να εκπαιδεύσουμε τον στρατό του Μάλι. Όντως υπάρχει μια επικάλυψη με τη μίσμα. Όμως, τα καθήκοντα της μίσμα σιγά σιγά τα αναλαμβάνει η ΕΚΟΑΣ, η Αφρικανική Ένωση και άλλοι δωρητές. Τώρα η προτεραιότητα της ευρωπαϊκής δύναμης είναι, μάλλον παραμένει η εκπαίδευση, το πρωτοτάγμα εκ 650 στρατιωτών του Μάλι εκπαιδεύτηκαν. Θα τελειώσουν την εκπαίδευσή τους σε λίγες εβδομάδες, δύο μήνες και μετά θα εκπαιδευτούν και άλλα τάγματα. Όπως είπα, δεν έχει αλλάξει κάτι στην μέθοδο εκπαίδευση της EUTM. Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή λοιπόν σε στρατιωτικέ δραστηριότητε, ούτε συμμετοχή σε άλλε ε, και πολύ μάλλον σε πολεμικέ δραστηριότητε. Όσον αφορά την ΕΚΟΒΑΣ και την Αφρικανική Ένωση, μετά από αυτήν την ε, μεταβατική περίοδο, ο ρόλος της ΕΚΟΒΑΣ θα είναι περίπου περισσότερο μάλλον ε, υποστήριξη της συμφιλίωσης, παρακολούθηση των εξελίξεων. Ακούγονται διάφορα τώρα για την διαδικασία συμφιλίωσης και δύο όσον αφορά τη διάσταση αποψε μεταξύ Μαυρετανίας, Νίγηρα, Αλγερίας από τη μια μεριά ως την άλλη άκρη του φάσματος. που πρεσβεύει μια πιο μειομορφή μεταχείριση του Βορρά. Δεν είναι τα πράγματα λοιπόν τόσο απλά όσο θα ήθελε να πιστεύει κανείς. Η Αφρικανική Ένωση επίσης παραμένει επιτόπου, σταθερά προσιλωμένη. Ο Πιερ Μπογιόγια, ο εκπρόσωπός της, ε, διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα. Μαζί με άλλους ειδικούς επεσταλμένους, όπως ο Μισελ Ρεβεράν Ντεμοντά, εκπρόσωπος των Ηνωμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται περισσότερο συντονισμός η ομάδα που συνεδρίασε στον Πάμακο την περασμένη εβδομάδα παραμένει απαραίτητη. Είναι μεγάλη ομάδα βεβαίω. Το θέμα είναι ο συντονισμός να είναι επικεντρωμένος, εστιασμένος. Αυτό θα βελτιώσει, ελπίζω, τα αποτελέσματα της διαδικασίας και ελπίζω να απήντησα και στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, τρεις επιπλέον ερωτήσεις και σας ξαναδίνω το λόγο αυτής αμέσως. Καθώς και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης του Τσάντ να αποσύρει 2.000 στρατιώτες από το Μάλι, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν ανταρτοπόλεμο, και το οποίο απομειώνει την δύναμη λοιπόν της διεθνούς δύναμη επιτόπου. Το ερώτημα είναι ποιο θα συμμετάσχει λοιπόν στην αντιτρομοκρατική δράση και στην εκπαίδευση. Δεύτερον, ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά την προοπτική εκλογών σύμφωνα με τι ε, προβλέψει, δηλαδή πρώτο γύρος 1 Ιουλίου και δεύτερος γύρος 31 Ιουλίου, μετά από τις ε, εξελίξεις, τις πολιτικές και άλλες εξελίξει του τομέα της στην περιοχή. Και τι είδου τεχνική βοήθεια σκοπεύει να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου. Επίσης, ποια είναι η γνώμη σα για την Σύνοδο των Δωρητών που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες προγραμματίζουν για τα μέσα Μαΐου συγκεκριμένα όσον αφορά την μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και της διακυβέρνησης. Δίνω και πάλι τον λόγο στον κ. Σοντόιλ και εν συνεχεία στο Συμβούλιο. Κυρία Πρόεδρε, οι δηλώσεις του Πρόεδρου του Τσάντ επί της ουσίας ε, είναι όπως το είπατε και εσείς ε, αυτές τα στρατεύματα του Τσάντ δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε έναν ανταρτοπόλεμο γιατί εκεί προς τα εκεί εξελίσσεται η σύραξη ο ρόλος τους ε, δεν μπορεί να είναι αυτός ένας τακτικός στρατός όπως φαίνεται και από την Ιγυρία δεν μπορεί να λάβει τέτοιου είδους καθήκοντα Τώρα, ποιος θα αναλάβει την αντιτρομοκρατική δράση, υποστήριξη κλπ. Πιστεύω ότι πρόκειται για συνδυασμό των τελευταίων δυνάμεων που θα αφήσει η Γαλλία στην περιοχή μαζί με κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα επεκταθούν ταχύτερα από δυνάμεις της περιοχής προκειμένου Πρόσφατα οι χώρες αυτές συζήτησαν θέματα συντονισμού για τους σκοπούς της ασφάλειας και τρίτον με εξωτερική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας να εξετάζουμε κάποια σενάρια. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο της ε, ΚΕΠΑ. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές του Ιουλίου, η έποψή μας ε, που είναι και η γνώμη εν πολλής και της ομάδας που συνεδρίασε την Παρασκευή ότι χρειαζόμαστε μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση για να μπορέσει να προχωρήσει η, συμφωλή, η συμφιλίωση και ο διάλογος. Σε πώς έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουν οι εκλογές, να γίνουν ακριβώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ο πρόεδρος Τσουνκούν ωραία. Ναι, ναι, ναι. αυτό ακριβώς είπε και λέει συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες. Συνεχίζει να τη χάνει κανείς υποστήριξη και πρέπει αυτή την υποστήριξη να την συνεχίσουμε. Τώρα, τι είδους υποστήριξη παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Αυτό τους άλλους ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες. Μητρώα, εκλογέων και ούτω καθεξής, μεταξύ άλλων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ληφθεί μια θετική ε, απόφαση υπέρ μιας πλήρης, πλήρους αποστολής παρατηρητών. Κάτι άλλο, η διάσκεψη της 15ης ε, Μαΐου. Αυτό με ρωτήσατε και τι περιμένουμε, τι είδους αποφάσεις για τον τομέα της ασφάλειας. Εκτιμώ ότι ο ήδη δρομολογηθής διάλογος θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε τα γνωστά θέματα, οι χώρε της περιοχής ε, εννοώ, ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, αλλά θα διευρυθούν και κάποιες ε, δραστηριότητες που έχουμε ξεκινήσει και στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας. Και ενδεχομένω όλα αυτά θα συνδυαστούν και με μια διεύρυνση της UCAP για το ΣΕΧΕΛ, της ε, δύναμης που έχει ως βάση την EMA. Μπορεί επίση να δοθεί νέα εντολή και να επεκταθεί η εντολή αυτή για να καλύψει το Τσάντ και ίσως και άλλες χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Que... Ευχαριστώ πολύ. Από το Συμβούλιο. Υπάρχει κανείς που θέλει να λάβει το λόγο. Euh, Όχι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που αντιπροσώπευε ο κ. Τζον Ντόιλ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση των σκέψεών του. Και προχωρώ στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, αλληλευτικοί περιορισμοί και χωρικά ύδατα στη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων. Έχω την τιμή να είμαι εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή, για την έκθεση αυτή. Ε, για την γνωμοδότηση που πρέπει να εκδώσουμε τους ώστε να ε, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βεβαίως η αλληλεία είναι πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει θέσεις εργασίας, δίνει πρωτεΐνες στους πολίτες, αλλά επειδή λόγω της πολύ έντονης εκμετάλλευσης των τελευταίων ετών οι πόροι γίνονται όλο και πιο σπάνιοι και για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους πόρους, αυτούς τους ελευτικούς πόρους θα πρέπει να πάρουμε ορισμένα μέτρα βεβαίως δημιουργούνται ε, συγκρούσεις βεβαίως δημιουργούνται ε, ε, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στις αποκλειστικές αλλιευτικές ζώνες ε, οι διαφορές όμως αυτές που δημιουργούνται θα πρέπει να επιληθούν ε, και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δώσουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες οικονομική και τεχνική βοήθεια που τη χρειάζονται για να μπορέσουν να ελέγξουν και τη διάρκεια των, και την νομιμότητα των αλληλευτικών δραστηριοτήτων στη, στα χωρικά του ύδατα. Όπως ξέ, ξέρετε υπάρχουν από χώρες οι οποίες δεν έχουν ε, άλλοι δεν έχουν σκάφη ελέγχου οπότε δεν μπορούν να ελέγξουν τα αλλιευτικά σκάφη και το τι κάνουν αυτά καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε την κατάσταση και στη Μεσόγειο και στον Εύξηνο ο Πόντο ούτω ώστε να μπορέσουν να, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να έχουμε μια βιώσιμη αλία, και όχι υπερβολική, τόσο ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους ελευτικούς πόρους. Σας υπενθυμίζω, μάλλον, να δώσω τώρα το λόγο σε, όποιον τον θέλει, ουδής. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μονικ Παγιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για το σχέδιο γνωμοδότησης. Πράγματι, η, η ε, Κομισιόν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ε, για ορισμένες περιοχές ε, και για τα μικρά νησιωτικά η Οι αλευτικοί πόροι είτε στα ενωσιακά ύδατα είτε εκτός είναι <clears throat> πρέπει να διατηρηθούν και βεβαίως οι οποιασδήποτε συμφωνίες κάνουμε βασίζονται στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και στις, στα ε, στοιχεία που έχουμε είναι από τις βασικές μας αρχές αυτό να διατηρήσουμε τους πόρους αυτή είναι η βασική αλληλευτική μας πολιτική η οποία έχει ε, υιοθετηθεί και από το Συμβούλιο θέλουμε και στις τρίτες χώρες και στα είδατα των τρίτων χωρών να υπάρχει ε, να εφαρμόζονται μέτρα ούτως ώστε να καταπολεμείται η, η παράνομη αλία θέλουμε να διατηρήσουμε τους αλληλευτικούς πόρους, να προωθήσουμε τη βιοπικιλότητα για να μπορούμε να έχουμε όλοι ίση και δίκαιη πρόσβαση και ελεύθερη πρόσβαση στους α, γενετικούς πόρους, τους αλληλευτικούς. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο και προσπαθούμε να προωθήσουμε την κύρωση και επικύρωση της UNCLOS και των άλλων συμφωνιών για τους ελευτικούς πόρους και βεβαίως να ε, συμφωνήσουμε και για τις μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων. Ειδικά αυτό το τελευταίο θέμα δεν είναι αντικείμενο της ε, περιφερειακής ε, της οργάνωσης ε, περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλίας αλλά ε, θα μπορούσε να συνδεθεί διότι τελικά ε, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, οι υπεύθυνοι είναι οι αρχές των παράκτιων χωρών με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή και προσπαθούμε να πείσουμε να δρουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε αποκλειστικές ελευτικές ζώνες με έναν τρόπο που είναι συμβατός με αυτά που κάνουμε στην Ένωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθήσουμε και οικονομικά και τεχνικά αυτές τις παράκτιες χώρες για να προωθήσουν τα προγράμματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουν θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις δυνατότητες για τις χώρες αυτές να δράσουν σωστά θέλουμε να συνάψουμε ε, συμφωνίες αλλιευτικές ούτως ώστε να γίνονται να πει, ακολουθούνται οι σωστές πρακτικές γίνονται σωστοί έλεγχοι, εποπτεία και τα λοιπά από τις χώρες αυτές τώρα ειδικότερα για τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο θα ήθελα να σας, υπευθυν... να υπενθυμίσω και την συμφωνία που σχετίζεται με τη συλλογή δεδομένων το σχετικό πρόγραμμα όπου από εκεί και πέρα τα εμπλεκόμενα κράτη ε, συνεργάζονται για τη συλλογή δεδομένων και υπάρχει και βεβαίως και η περιφερειακή οργάνωση για τη Μεσόγειο στην οποία συμβάλλει σημαντικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον συγχρηματοδοτούμε πολλά έργα μαζί με την ΦΑΟ γιατί υπάρχουν προγράμματα ειδικά για τη Μεσόγειο τόσο ώστε να βελτιωθεί η συλλογή επιστημονικών δεδομένων. Και βεβαίως το ίδιο θα κάνουμε και στη νέα προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης ευχαριστεί ιδιαίτερα τον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα την Επίτροπο Αλίας για όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει για να προχωρήσουμε σε μια βιώσιμη ε, αλία. Βεβαίως οι συμφωνίες ηλιευτικές οι οποίες ε, συνήφθησαν πρόσφατα είναι καλύτερες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στις, ε, ε, συναντήσεις τριμερούς διαλόγου που θα λάβουν χώρα. Ελπίζουμε πραγματικά να οδηγηθούν οι συναντήσεις αυτές σε επιτυχία <clears throat> για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία λοιπόν για τους ε, τη συναντήσει αυτή του τριμερούς διαλόγου. Σας υπενθυμίζω ότι η κατάθεση τροπολογιών μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 28 Μαΐου. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης για το πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς και τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στο ωφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους το οποίο επισυνάπτει τη σύμβαση για την βιοπικιλότητα. Η συγκεκριά μας για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η Κατρίν Γκρέζ. τα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη σε σχέση με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη δίκαιη με ε, συμμετοχή στα ωφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους θα συζητηθούν ε, από κοινού. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον έχει ε, συντάξει δύο γνωμοδοτήσεις για τις ε, εκθέσεις αυτές. μία αφορά το πρωτόκολλο της Ναγκόγια και το άλλο αφορά ένα σχέδιο κανονισμού για την υλοποίηση του πρωτόκολλου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς χρονοτριβή, λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέζ για να μας παρουσιάσει αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να επανέλθω στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα σε αυτήν την Επιτροπή και στην Ολομέλεια για την έκθεση πρωτοβουλίας που παρουσίασε για τη βιοπειρατεία που κατά την ε, άποψή μου πραγματικά έσπασε τα ταμπού που είχαμε για τη βιοπειρατεία η βιοπικιλότητα στον κόσμο ε, τελικά είναι ε, κάτι κοινό, μειώνεται μέρα με τη μέρα και ε, ξέρετε, ειδικά σε αυτή την Επιτροπή έχουμε μία ευθύνη προκειμένου να μην κλείσουμε τα μάτια μπροστά στις καταστροφικές συνέπειες της μείωσης της βιοπικιλότητας για τους τοπικούς πληθυσμούς παγκοσμίους. Θα ήθελα να πω πως αυτή η απώλεια βιοποικιλότητας και η καταπολέμηση αυτής της απώλειας βιοποικιλότητας δεν είναι μια επιλογή. Η βιοποικιλότητα πράγματι είναι κάτι ζωτικό. Και αφενός έχουμε ε, προμηθευτές γενετικών πόρων ε, και προφανώς έχουμε και τους κατόχους των παραδοσιακών γνώσεων που και στις δύο περιπτώσεις ε, στην πλειονότητά τους προέρχονται από τα ανεπτυσσόμενες χώρες. Η βιοπικιλότητα επίσης και η ποικιλότητα αυτής της ε, βιοπικιλότητας ε, συχνά ε, κοιτάει στις λεγόμενες χώρες του Νότου. Επίσης, ξέρουμε το 70% του πληθυσμού που βρίσκεται σε δίνη κατάσταση κατέχουν ε, την ε, βιοπικιλότητα και είναι πολύ σημαντική αυτή η βιοπικιλότητα για αυτούς. Ε, το νερό είναι μια πηγή ε, εσόδων επίσης και είναι και σημαντική για το κλίμα. Επομένως, η υποβάθμιση του κλίματος ζημιώνει ιδιαίτερα την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία την, ενός μεγάλου μέρους ειδών και Επίση, τίθεται και σε κίνδυνο η επιστηστική ασφάλεια και η ανάπτυξη μιας αηφόρου γεωργίας σε πολλές ερωτευσόμενες χώρες. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έκανε μια νομοθετική πρόταση για να θέσει σε εφαρμογή το πρωτόκολλο της Ναγκόγια και αυτό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον γιατί αυτό το πρωτόκολλο είναι το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τη βιοπειρατεία. Να σας υπενθυμίσω, η Σύμβαση για την Βιοπικιλότητα, η CBD, και προφανώς το πρωτόκολλο της Ναγκόγια, και εδώ θα παραθέσω κείμενο ε, υποθέτουν την προηγούμενη συγκατάθεση των χωρών προέλευσης ή των τοπικών και γηγενών κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με τους γενετικούς πόρους και μέσα με αυτές πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες, για, κατάλληλοι όροι για ε, τις ε, συμφωνίες, διαδικασίες συνένεσης μετά από ενημέρωση και μηδέν συμφωνηθέντες όροι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρωτόκολλο της Ναγκόγια που βασίζεται σε τρεις ε, πυλώνες. Το πρώτο είναι η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους ε, που προφανώς ε, δεν το προσεγγίζει το θέμα αυτό η πρόταση της Κομισιόν γιατί έχει να κάνει με την κυριαρχία των διάφορων χωρών. Το δεύτερο πυλώνας που είναι ο καταμπορισμός των ωφελών που προκύπτουν από τους ε, πόρους. Ασχολείται με το θέμα αυτό η Κομισιόν, αλλά όχι αρκετά κατά την γνώμη μου. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ο σεβασμός των κανόνων από τους χρήστες και οι κυρώσεις. Αυτά τα σχολιάζει η Κομισιόν στην πρότασή της. Επίσης, διαπιστώνω ότι η πρόταση που μας υποβληθήκε προσανατολίζεται πολύ περισσότερο προς ε, το συμφέροντα των χωρών χρηστών παρά των χωρών προμηθευτών. Αυτό δεν με εκπλήσει. Ε, δηλαδή αφορά ε, εδώ περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρες το θέμα αυτό και όπως κάναμε και με την έκθεση πρωτοβουλίας εδώ έχουμε για μια ακόμη φορά ευθύνη να υπερασπίσουμε τη συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης και να αποκαταστήσουμε μία ορθή ισορροπία μεταξύ των προμηθευτών και των χρηστών. Αν ε, μου επιτρέπετε να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα μπω στις λεπτομέρειες των όσων προτείνονται. Η αρχή της ε, δέουσας επιμέλειας που αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν. Δηλαδή, το ότι υποχρεούνται οι χρήστες να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, τα απαραίτητα διαβήματα, αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να το συναδεύσουμε και με την αρχή της απαγόρευσης της βιοπειρατείας και να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση και τη χρήση γενετικών πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα. Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να καλύπτει και τις νέες χρήσεις των γενετικών πόρων ε, και των σχετικών γνώσεων. Έχουμε πάρα πολλού γενετικού πόρου, ε, του γνωρίζουμε, υπάρχουν στι συλλογέ και δεν καλύπτονται από τι προτάσει κανονισμού. Θα πρέπει λοιπόν το πρωτόκολλο τη Ναγκόγια να εφαρμόζεται και για κάθε νέα χρήση γενετικών πόρων. Τρίτον, μια ιδέα που μου φαίνεται πολύ σημαντική είναι η εξή. Μέχρι να φτάσουμε στον παγκόσμιο πολυμερή μηχανισμό, κάτι που είναι πολύ φιλόδοξο, να μπορέσουμε να, χρησιμοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης μία βάση για το είναι κατανομή των ωφελών. Παραδείγματο χάρη, αν σκεφτούμε τους πόρους της ανοιχτή θάλασσας ή τους ιστορικούς, όπως λέγονται, πόρους. Ε, είναι ε, δυνατόν να βρούμε την προλευσή τους. Έτσι λοιπόν, ε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συλλέξουμε τα ωφέλη σε μια οπτική διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Τελευταίο σημείο, τέταρτο σημείο, βελτίωση της αλυσίδα της χρήσης γενετικών πόρων και των σχετικών γνώσεων. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να επιτρέψουμε την ανεχνευσιμότητα και την ασφάλεια δικαίου για τους χρήστες. Πρέπει λοιπόν να θεθεί σε εφαρμογή ο έλεγχος και να γίνουν και επαληθεύσεις, κάτι που φαίνεται ουσιαστικό και φτάνω στα συμπεράσματα. Είναι απολύτως σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των αυτοχθόνων ε, γίνονται σεβαστά καθ' όλη την ελισίδα της χρήσης, προκειμένου να υπάρχει πραγματικός επιμερισμός και ισότιμος επιμερισμός των ωφελών. Όχι μόνο οικονομικός, αλλά και με ένα σύστημα που να είναι πιο σαφές, πιο αποτελεσματικό και να μας επιτρέπει να καταπολεμήσουμε το διοικητικό άχθος. Η υλοποίηση του πρωτοκολλού αυτού της Ναγκόγια, κατά την άποψή μου, θα πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψη τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο όσο τις αναπτυγμένες χώρες. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να εκπονηθεί μια νομοθεσία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την κατανομή των ωφελών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Και αυτό σημαίνει να ενισχύσουν σημαντικά οι ικανότητες σε νομικό και θεσμικό επίπεδο στις χώρες αυτές. Ελπίζω να μου μακρηγόρησα πολύ. Κατανοήσετε ποια είναι η φιλοσοφία που αναπτύσσω εδώ. Ακολουθεί τα όσα συζητήσαμε και τα όσα είχαμε συμφωνήσει όταν εκπονήθηκε η έκθεση πρωτοβουλίας για τη βιοπειρατεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Οι βουλευτές το λόγο το επιθυμούν. Παρακαλώ, κύριο Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για την έκθεσή της. Είναι μια ισορροπημένη και πολύ καλή ε, έκθεση γνωμοδότησης. Ε, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και ήταν ε, πραγματικά καιρός για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να το ε, υιοθετήσει, να το περάσει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και να αρχίσει η εφαρμογή του. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε προφανώς το 1992 στην, στην, στην συνάντηση του Ρίο ε, αλλά ήταν μόλις το, στην Αγκόγια το 2010 που πραγματικά ε, φτάσαμε στην υπογραφή του πρωτοκόλου που τι κάνει, κάνει το αυτονόητο. Βάζει stop σε μια παράνομη δραστηριότητα στην βιοπειρατεία. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια ε, αυτό που κάνει είναι να αποδίδει, να υποχρεώνει τις εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, πόρους, βιολογικούς πόρους, να έχουν, πρώτη, να έχουν έγκριση από τις τοπικές ε, κοινότητες, είναι κράτος ή, ή άλλες, ε, ή άλλες διαβαθμίσεις ε, τοπικής αυτοδιοίκησης, να, έχουν, ε, να μοιράζονται τα ωφέλη με, αυτήν την, ε, με αυτές τις κοινότητες από τις οποίες προέρχεται η, αυτός ο πόρος. Είναι ένας πρώτος, ε, ένα πρώτο στάδιο, μια πρώτη προσπάθεια να μπει ένα φρένο στην βιοπειρατεία. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαπραγματεύση στην Αγκόγια ε, είχε για μεγάλο διάστημα αρνητική στάση στο πρωτόκολλο, με πάρα βάζοντας πάρα πολλά εμπόδια. Τα, με την πίεση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι βελτιώθηκε, αλλά και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρωτόκολλο που μπορεί να μην είναι τέλειο κινείται προς σωστή κατεύθυνση και συμφωνώ και με τις προτάσεις της ε, εισηγήτριας και στην έκθεση γνωμοδότησης. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ε, στην έκθεση αυτής της γνωμοδότησης και στην, ε, υιοθέτηση του πρωτοκόλλου την υπογραφή του πρωτοκόλου επίσημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο Γκουσάλη ή στον κύριο Βασίλη Κουτσουρή. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω στη συζήτηση της σε ό,τι φορά το πρωτόκολλο της Ναγκόγια και την εφαρμογή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε ε, κανόνες συμμόρφωσης για τους ε, χρήστες ε, και για την επιμερισμό των ωφελών με τις χώρες προμηθευτές. Η Κομισιόν μετά από διαβουλεύσεις με όλα τα διαφορεμένα μέρη και μετά από μία μελέτη δικτύπου εκτεταμένη όπου συζητήθηκαν όλες τις δυνατότητες παρουσίασε την πρότασή της η Κομισιόν. Η δική μας πρόταση θέτει κανόνες για του χρήστες και προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των προμηθευτών και των χρηστών. Χωρίς αποτελεσματική ασυμόρφωση των χρηστών, η κυριαρχία των αλδοπών χωρών δεν μπορεί να γίνει σεβαστή. Η πρότασή μας προσφέρει μια αποτελεσματική λύση για την πρόσβαση και την κατανομή των ωφελών που είναι επίσης ε, αξιόπιστη για τους άλλους εταίρους μα και μπορεί να διευκολύνει τις μελλοντικές συμφωνίες ε, ή ε, ο πολλαπλασιασμό των συμβάσεων ε, θα επιφέρει περισσότερα ωφέλη που θα μοιραστούμε με τις υπόλοιπες χώρες. ο κανονισμός καλύπτει τους γενετικούς σπόρους που έχουν τεθεί αφού τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο της Ναγκόγια στην Ένωση. Αυτό σέβεται το πρωτόκολλο της Ναγκόγια και ε, θέτει ασφάλεια δικαίου για τους χρήστες να επενδύσουν ε, και ε, αυτό βάσει των γενετικών πόρων. Επίσης έχουμε υποχρέωση δέωσης επιμέλειας ως το κύριο μέσο για τη συμμόρφωση των χρηστών. Δεν πιστεύουμε και δεν υποστηρίζουμε την ιδέα να είσαι μια απαγόρευση για τη συμμόρφωση των χρηστών. Μια απαγόρευση θα ε, αφαιρούσε κίνητρα από τους ε, περαιτέρω χρήστες ε, για να γίνει έρευνα και ανάπτυξη βάσει των γενετικών πόρων θα χρήσονταν ε, ομοιόμορφα πρότυπα για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, κάτι που τώρα δεν ισχύει. Επίσης θα πετούσε ορισμό της ε, παράνομης χρήσης ή της ορισμοί που θα πρέπει να εκπονηθούν καταρχήν σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να παραπέμψω στη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της υπόθεσης νομικών θεμάτων, ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής δικτυσίας ε, και του Ιανουαρίου 2013, όπου επίσης αναφερόταν και ανάγκη για διευκρίνηση και επαγίωση των ορισμών αυτών. Ο κανονισμός θέτει ένα σύστημα checkpoints ως στην αρχή και στην, ε, στο τέλος της αλυσίδας των χρηστών που απαντά ε, στις απαιτήσει του άρθρου 17 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Δεν πιστεύουμε ότι περισσότερα checkpoint και υποχρεώσει για τους χρήστες θα συνεισφέρουν σε καλύτερη εφαρμογή των υποχρεώσεων των χρηστών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους ελέγχους επί της που πρέπει να κάνουν το κράτη-μέλη δύναμη του άρθρου 9 μέσα στα όρια του πρωτοκολλού της Ναγκόγια η πρότασή μας σέβεται και προωθεί τα δικαιώματα των αυτοχθόνων σε σχέση με την παραδοσιακή γνώση και τους γενετικούς πόρους. Η πρότασή μας δεν υπερασπίζει τη δημιουργία ενός παγκοσμίου μηχανισμού κατανομής των ωφελών περιμένοντας τα μέρη της Ναγκόγια να καταλήξουν σε παγκοσμία λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενεργή στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της διάσκεψης των μέρων τη CBD, συγγνώμη, ε, τα μέρη του πρωτοκολλού της Ναγκόγια όταν τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο θα πρέπει να καθορίσουν τους ε, ανάγκες και τους τρόπους αυτού του πολυμερούς μηχανισμού καλύπτοντας μία σειρά περιπτώσεων ε, όπου δεν μπορεί να αποκτηθεί δυνατότητα επιλογής του ότι μας αρέσει παράλληλα. Παράλληλες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα για, με την Άγγλος για μία εφαρμοστική συμφωνία με την Άγκλο σε πέρα της εθνικής δικαιοδοσίας. Πιστεύουμε ότι δεν ε, ε, θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτές ε, τις την αναζήτηση επικοσμίων λύσεων. Αν έχω χρόνο, θα μπω σε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με την πρόταση. Μπορώ. Ευχαριστώ σε για συγκεκριμένες πτυχές ε, της, ε, των τροπολογιών. Εμείς θεωρούμε το εξή. Σχέση με το άρθρο 2, ο κανονισμός ε, δεν καλύπτει τους γενετικούς μόρους σε τομείς πέρα της εθνικής δικαιοδοσίας και συνάδει με τα άρθρο 15 της CBD και 3 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Η πρόταση για το άρθρο 5 για πρόσθετες δραστηριότητες ε, των συλλογών είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές προς το κόστος. Πιστεύουμε ότι θα αποτρέψει τις συλλογές από το να γίνουν trust collections. Για το άρθρο 7 στην ε, ε, πολυπλασιασμό των checkpoints, αυτό δεν προσθέτει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος. Άρθρο 8, βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι τις πρακτικές δυνάμει του άρθρου 8 είναι εργαλεία εφαρμογής ε, που διευκολύνουν τη συμμόρφωση του χρήστη. Οι ιδέες που προτείνονται υπό αυτό το άρθρο μπορεί ε, να... να εφαρμοστούν στο μέλλον όταν συζητήσουμε το άρθρο 14 για τα συμπληρωματικά μέτρα. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο τώρα στην κυρία Γκρέζ για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη σημείωσα τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει μια κάποια ισορροπία μεταξύ προμηθευτών και χρηστών αλλά σημείωσα επίσης και ορισμένα σημεία όπου δεν υπάρχει συμφωνία και που πρέπει, στα οποία ακόμη πρέπει να δουλέψουμε. Ε, πιστεύω πραγματικά ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας μέσα στο ίδιο πνεύμα που μας ανέπνευσε και για τη βιοπειρατεία. Πρόεδρος, Λοιπόν, οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 30 Απριλίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 28 Μαΐου. Θα ήθελα με την ε, ε, άδεια της εισηγήτριας να αντιστρέψω τη σειρά της ημερήσιας διώτηξης για να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω τον Πρωθυπουργό της Κεντροαφρικανικής Ένωσης Όπως σας είπα στην αρχή της συνεδρίασής μας, η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι ασταθής και ανησυχητική. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να συζητήσουμε ακριβώς αυτή την κατάσταση, όπως και τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της χώρας, ε, που είναι θύμα των που φυσικών της πόρων έχει πολλούς φυσικούς πόρους η χώρα αυτή αλλά παραμένει πάρα πολύ φτωχή είναι θύμα της μοίρας της έννοια μετά από τις ε, ε, διαμάχες της Περσινές και της αρχής της χρονιάς τελικά ε, ξεκίνησαν οι εργασίες για μια συμφωνία στη Λιμπρβιλ είστε επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης και ο τέος πρόεδρος της χώρας ο κύριος Μπουασισέ ε, το τότε απομακρύνθηκε στις 24 Μαρτίου. Ο κύριος Τσότο Ντίντια ε, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας που από καθήλωση τρόπων την προηγούμενο πρόεδρο ε, αποφάσισε ε, δήλωσε ότι θα κυβερνήσει μέσω προεδρικών διαταγμάτων για τρία χρόνια και μετά θα γίνουν εκλογές. Ο κύριος Τσοτοντία βεβαίω μετά από τις αντιρρήσεις που υπήρχαν σας, σας ζήτησε ξανά να φτιάξετε μια μεταβατική κυβέρνηση και ο, ε, ε, υπάρχει, δημιουργήθηκε ένα συμβούλιο μεταβατικό το οποίο όρισε τον κύριο Τσοτοντία ε, ως πρόεδρο για 18 μήνες οι εκλογές ε, στις οποίες αναφερόταν ο, στις οποίες δεν θα λάβουν μέρος ούτε ο κύριος Τσότο Ντία ούτε ο, τα μέλη της κυβέρνησής του εντός εισαγωγικών θα λάβουν χώρα αργότερα και ε, το Συμβούλιο θα ετοιμάσει ένα σχέδιο συντάγματος το οποίο, για το οποίο θα γίνει δημοψήφισμα και αν ε, και βεβαίως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καινούργια διαδικασία μεταβατική αδυστυχώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρεμία έχει επανέλθει στην πρωτεύουσα Μπαγκουή αντιθέτως την περασμένη εβδομάδα ε, έγιναν ε, συγκρούσεις οι οποίες είχαν και θύματα και ζητήσατε κύριε Πρωθυπουργέ τη βοήθεια διεθνών στρατευμάτων για να επανέλθει η τάξη Υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας στην περιοχή και εκείνο που τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ή όλοι μαζί είναι ότι η διαδικασία η μεταβατική θα είναι μια διαδικασία στην οποία να συμμετέχουν όλοι, όλοι τα μέτρα τα οποία παίρνονται βάσει θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά και οι βασικές αρχές θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Όπως το είπατε και ο ίδιος υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις. Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας και μπορούμε να συζητήσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις με εσάς προσωπικά. Έχετε το λόγο κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με δεχθείτε εδώ και εμένα και την αντιπροσωπεία μου για να σας παρουσιάσουμε σύντομα την κατάσταση στη χώρα μας. Το, η σύντομη παρουσίαση που κάνατε εσείς πράγματι δίνει ορισμένα στοιχεία για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, στην χώρα μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνω κι εγώ μια ιστορική ανασκόπηση ε, του τι συμβαίνει σε μας. Η χώρα μου είναι ενδυνάμει πλούσια. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια ε, υπόκειται ε, αντιμετωπίζει προβλήματα ε, ανταρσιών, πραξικοπημάτων κτλ. Από τις 24 Μαρτίου του 2013 μια ομάδα ανταρτών ε, έχει στα χέρια της την εξουσία στη χώρα μας και αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, προκλήσεις πολιτικές και συνταγματικές θέλουμε να επανέλθουμε σε μια συνταγματικά ήρεμη κατάσταση ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα εντός 18 μηνών αν είναι δυνατόν και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα προσχέδιο συντάγματος το οποίο θα παρουσιαστεί στο λαό γιατί προβλέπεται δημοψήφισμα ε, το όργανο που θα ετοιμάσει το προσχέδιο αυτό είναι ένα όργανο, είναι το Εθνικό ε, Συμβούλιο Μεταβατικό Συμβούλιο το οποίο ε, δημιουργήθηκε ε, μετά την ε, έκτακτη συνάντηση στις 3 Απριλίου και το οποίο Συμβούλιο νομιμοποιεί τρόπον την αντικατάσταση που υπάρχει στη χώρα μου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση μεταβατική και προ προς την ομαλοποίηση της κατάστασης αν θέλετε υπάρχουν πολλές προκλήσεις υπάρχει ανθρωπιστική ε, πρόκληση γιατί στη χώρα μου μετά από τις ένοπλες που έγιναν τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε η χώρα μου βρίσκεται σε άσκημη ανθρωπιστική κατάσταση ε, έγιναν λαιλασίες, έγιναν σφαγές, έγιναν ε, ε διώξεις που κατέληξαν τελικά στα 1,5 εκατομμύριο άτομα να έχουν εκδιωχθεί από το χώρο τους. Είναι πολύ μεγάλο το, πολύ μεγάλο το νούμερο αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό μιλάμε για ε, πραγμα... ανθρωπιστική κρίση, ανθρωπιστική τραγωδία. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και προκλήσεις οικονομικές και κοινωνικές, διότι ο κοινωνικός ιστός διαλύθηκε, η οικονομία διαλύθηκε, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει χωροφυλακή, δεν υπάρχει αστυνομία και όπως είπατε επικρατεί αταξία, αναρχία στη χώρα μου διότι το κράτος ως οργανωμένη εξουσία δεν υφίσταται πλέον. Δεν υπάρχει στρατός όπως σας είπα, δεν υπάρχει ενοποιημένη στρατιωτική δύναμη αν θέλετε που μπορούμε να, η οποία μπορεί να δράσει. Βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς πραγματικής αναρχίας. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στη χώρα μου και χαιρόμαστε που μπορούμε, που βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε αυτή την δυστυχή πραγματικότητα ε, στην οποία, την οποία βιώνουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ. Ο λόγος τους βουλευτές, ο κ. Λουί Μισελ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζήτησαν να παρέμβω διότι ο Πρωθυπουργό βεβαίω δεν μπορεί ίδιος να μιλήσει για τα προσόντα που τον ορίζει η διεθνή κοινότητα. Ο Γενικό Γραμματέα τη Γαλλοφωνία στι 3 ε, Απριλίου ήμουν στην Τζαμένα όπου έγινε η δεύτερη έκτακτη συνδιάσκεψη Λαμβάνω λοιπόν τον λόγο για να πω ότι ο Πρωθυπουργό δεν ήταν ούτε είναι εκπρόσωπος της ΣΥΝΤΕΚΑ. Όμως ομοφόνος αναρωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Κέντρο Δημοκρατία ως ε, ο άνθρωπο ο οποίο θα σώσει την κατάσταση. Εμεί ε, οφείλουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του, το κύρος του. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Αναγνωρίζεται επίσης ομοφόνος από όλη την ε, διεθνή κοινότητα, από την Αφρικανική Ένωση ως τα ένα Έθνη, μεταξύ άλλων ε, από την Γαλλοφωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζεται λοιπόν από όλους, διδραμάτισε ρόλο κατευνασμού και επίσης ε, επηρεάζει τον αυτοποκαλυμμένο πρόεδρο είναι ο Πρωθυπουργό, ο οποίος ε, έθεσε τα πρώτα, έκανε τα πρώτα βήματα σε έναν εναρετό κύκλο για καλύτερες μέρες στη χώρα. Δυστυχώς, η Σελικά εκπροσωπείται από ανθρώπους ε, απρόβλεπτου. Η απόφαση της Τζαμένα να ενισχύσουμε τα στρατεύματα από χώρε τη περιοχής, ήταν καλή απόφαση, για να ανακουφίσουμε λίγο τους πολίτες της περιοχής. Αυτό το εγχείρημα πρέπει να τον ισχύσουμε περαιτέρω. Το θέμα της χρηματοδότηση όμω παραμένει ανοιχτό. Η κεντροαφρικανική δημοκρατία, ό,τι υπομένει από αυτήν, είναι κράτος με άδεια ταμεία με κίνδυνο βεβαίω κοινωνική έκρηξη. Αν συνδυάσετε την κατάσταση με την βία στους δρόμους, με τις απόπειρε, τις στοχευμένες απόπειρες, τον κίνδυνο θρησκευτικών διαμαχών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν δεν επιληθεί και το οικονομικό πρόβλημα θα οδηγηθούμε σαφώς σε έκρηξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Πρωθυπουργό. Έλαβα λοιπόν, επαναλαμβάνω τον λόγο για να θυμίσω σε ποιο βαθμό η διεθνή κοινότητα υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται για έναν άνθρωπο εξαιρετικά μετριοπαθή, ε, πρόκειται για έναν άνθρωπο χωρίς προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίε, Ξέρουμε άλλωστε ότι ούτε ο πρόεδρο, ούτε ο θα έχουν την δυνατότητα να είναι υποψήφοι στις εκλογές, τις προεδρικές ή τις κοινοβουλευτικές. Οπότε από εδώ και πέρα πρέπει ο χάρτης πορείας να αποκριστελωθεί. Ε, βέβαια υπάρχει αυτός ο χάρτης, εδώ και τρεις μέρες ε, προκρίθηκε στην ε, Τζεμένα. το Υπουργικό Συμβούλιο βεβαίω πρέπει να γίνει πολύ πιο αντιπροσωπευτικό. Χρειάζεται ένας ανασχηματισμός και μια μεταβατική ε, βουλή, η οποία θα μπορέσει να νομοθετήσει, θα αντικραστήσει τη σημερινή βουλή που έχει διελθεί και μια συντακτική βουλή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και τέλος, ε, για να μείνουμε ακριγόρο, Εννοείται ότι όλοι είμαστε υπέρ της επιστροφής στην συνταγματική τάξη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όμως το εκλεχθισόμενο κοινοβούλιο θα αποτελείται από 100 μέλη της πλειοψηφίας. Οι παρατηρητές είχαν διαπιστώσει θέματα νομιμότητας των εκλογών. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, ότι υπήρχε πρόβλημα. Και τέλος δεν άκουσα κανέναν από αυτούς με τους οποίους μίλησα τουλάχιστον και μίλησα με πολλούς πρέπει να ξέρετε. Δεν άκουσα, επαναλαμβάνω, κανέναν να παραπονείται για την έξοδο του Πρόεδρου. Είναι σημαντικό αυτό να το πω, γιατί είναι και δική μας, αν θέλετε, επιθυμία και είναι και μια έκκληση που απευθύνει αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργό μα που δέχτηκε την πρόσκλησή μα θα συνθεί με διάφορε προσωπικότητε στην Ευρώπη. Τον καλό να μα βοηθήσει και θα τον υποστηρίξουμε για να αντιμετωπίσει, να αντεπεξέλθει στην, στις προκλήσεις και στις προσδοκίες ενός λαού ο οποίος ε, υποφέρει. Βλέπει ότι υπάρχουν προοπτικές, ε, πόροι, έσοδα ε, και δυστυχώς αυτοί οι πόροι να μην αξιοποιούνται εδώ και πολύ καιρό για το καλό του λαού της χώρας. Ο κ. Σίγκα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί με την προπόθεση ότι θα βοηθήσει η διεθνή κοινότητα. Δεν χρειάζεται βοήθεια μόνο από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συμπρόεδρο της ε, κοινοβουλευτικής, ε, της μεικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρονακέ και Γενικό Γραμματέα της και Κυρία Σαρκεντίνη. Κυρία Πρόεδρε, εάν χρειάζεται μετάφραση ο Πρωθυπουργός, περιμένω για λίγο, πολύ ωραία, για να βάλει τα ακουστικά του. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ που ήρθατε στην εισαγωγή της Πρόεδρου. Ακούγομαι. Να περιμένω. Με ακούτε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Η εισαγωγή της Πρόεδρου μας. Η Πρόεδρος ε, χρησιμοποίησε την κατάσταση αναφέροντας την, την κατάρα των πόρων. Ε, λοιπόν, ήθελα να πω ότι χαίρομαι που είστε εδώ και χάρηκα που σας άκουσα να λέτε ότι χώρα αυτή τη στιγμή, στη χώρα αυτή τη στιγμή βασιλεύει ενέργεια και ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Εν τούτης, η χώρα δεν ήταν και φάρος της δημοκρατίας ε, πριν το πρόσφατο πραξικόπημα. Ο πρόεδρος Μποζής κυβέρνησε επί 10 χρόνια. Τα δέκα αυτά χρόνια έβγαλε πολλά από το εμπόριο διαμαντιών, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας μιλήσετε για το πώς βλέπετε εσείς τις ευκαιρίες τεθροποίησης της χώρας. Τι χρειάζεται από εμάς, αλλά και τι μπορεί να κάνει η ελίτ της χώρας ώστε αυτή η κατάρα να πάρει τέλος. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει ως Πότε θα δούμε εκλογέ, πότε θα ανανεωθεί, πότε θα αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα. Και τρίτον, διάβασα δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και Υπουργού Αμήνη τη Νότια Αφρικής και δικές δηλώσει δηλώσει σχετικά με την επιστροφή νοτιοαφρικανών στρατιωτών στην περιοχή. Ήμουν στην Νότια Αφρική πριν από λίγο καιρό, όταν ο Υπουργό ε, Αμήνη εξηγούσε τι έκαναν, ποιο ήταν ο ρόλο των νοτιοαφρικανών στρατιωτών στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ε, εγώ ρωτώ ότι και πάλι ε, αυτό δεν είναι σαφέ. Προστατεύουν μήπω μόνο Πόρου που ανήκουν στην Νοτιοφρική, οι τη Νότια που όμω όλα μα επιστρέφουν στη γνωστή κατάρα των πόρων, για την οποία μιλήσαμε λίγο πριν. Θα ήθελα να μα μιλήσετε για όλα αυτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Αν κάποιο ε, θέλει να πάρει το λόγο τη Επιτροπή, κανεί. ούτε κάποιο από την υπηρεσία εξωτερική δράση. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Πρωθυπουργό για να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους βουλευτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Βλέπω ότι γνωρίζετε την πραγματικότητα της Κεντρικής αρχής, ε, γιατί μιλήσατε για τη δεκαετία του Μποζής, ε, όπου είχαμε μια λαϊλασία ε, των πόρων της χώρας μας και συγκεκριμένα των διαμαντίων, γιατί ο Μποζής πράγματι πλούτησε πάρα πολύ λαϊλατώντας τον πλούτο μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιμένουμε μια οικονομική βοήθεια στην πραγματικότητα, γιατί όπως ήδη είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος οικονομικός εταίρος της ε, χώρας μου, της ε, Δημοκρατίας και της Αφρικής. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, αν ε, υπήρξε ε, ανατροπή της τάξης θα μπορούσε να σταματήσει την υλοποίηση αυτών των έργων. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοια αναστολή που θα ζημιώσει τα συμφέροντα του πληθυσμού που ήδη υποφέρει πάρα πολύ. Δεύτερον, για την αποκατάσταση της σταθερότητας ε, της χώρας. Ήδη έχουμε αυξήσει ε, τα στρατεύματα της ΦΟΜΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση των δυνάμεων της ε, οικονομικής κοινότητας στην δύναμη της ΦΟΜΑΚ, που είναι η δύναμη της Κεντρικής Αφρικής, προκειμένου να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει να παρέχει χρηματοδότηση για τα στρατεύματα. Και από 700 θα φτάσουμε στους 2.000 άντρες στα στρατεύματα αυτά. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει ούτε σέντς ε, ε, στα κρατικά ταμεία. Δεν έχουν καταβληθεί οι μισθοί ούτε για τον Μάρτιο ούτε για τον Απρίλιο. Ήδη έχουμε 22 Απριλίου. Έτσι λοιπόν μία επίγουσα βοήθεια θα μπορούσε να μας επιτρέψει να καλύψουμε τα κατεπήγοντα γιατί τα στοιχεία που προκαλούν ε, αναταραχές στην πρωτεύουσα είναι τα στοιχεία του ΣΕΛΕΚΑ. Και για να τις αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να ξοδέψουμε πάρα πολύ χρήματα και τώρα το κράτος δεν τα έχει τα χρήματα αυτά, θα πρέπει να το στρέψουμε και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα ε, ότι θα έχουν συσταθεί τα κατάλληλα όργανα για τη μετάβαση. Η κυβέρνηση δεν έχει τα μέσα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτές ε, τις τεράστιες υποχρεώσεις και γι' αυτό πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τη βοηθήσει για να ρυθμίσει αυτές τις δυσκολίες. Επίσης, να επανέλθω στο ότι οι αντάρτες κατέστρεψαν όλα τα κτίρια τα διοικητικά. Δεν ε, υπάρχουν πλέον υπολογιστέ, ε, ούτε καρέκλες, ούτε τραπέζια. Επομένως, δεν υπάρχει καν η δημόσια διοίκηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τα μέσα στο εγγύς μέλλον να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σκεφτόμαστε ότι μια οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ευπρόσδεκτη. Δηλαδή να έχουμε μια κατεπίγουσα δημοσιονομική βοήθεια. Αυτό για την πρώτη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στρατεύματα της Νοτιοαφρικής, ο πρόεδρος ε, Ζούμα κατά την έκτακτη σύνοδο κορφής στις 18 Απριλίου ζήτησε να συναντηθεί με την ε, κυβέρνηση της Κεντρικής Αφρικής και μία αποστολή θα μεταβεί στην, ε, στην Κεντρική Αφρική για να συζητηθεί η συνεργασία με το δύο χωρών, γιατί η συνεργασία μεταξύ Κεντρική Αφρικής και Νότια Αφρικής μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν από προσωπικά συμφέροντα που δεν είχαν καμία σχέση με τα συμφέροντα των κρατών. Γι' αυτό η αποστολή που θα μεταβεί στην Νότια Αφρική θα έχει ως καθήκον να αποσαφηνίσει τη φύση των σχέσεων που υπήρχαν μέχρι σήμερα μεταξύ του Μποζίσε προσωπικά και κάποιων ε, άλλων που εκπροσωπούσαν προσωπικά συμφέροντα από την Νότια Αφρική. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Merci. ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μας απομένει παρά να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και πολλή ενέργεια για να υλοποιήσετε αυτά τα πολύ σημαντικά καθήκοντα. Και επίσης να ελπίσουμε ότι θα ακουστούν οι εκκλήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Και ευχαριστώ και όλους τους αξιότιμους κυρίους βουλευτές. Να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερησία διάταξη. καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη, μια βιοοικονομία για την Ευρώπη. Η κυρία Λέβιν έχει συντάξει ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την Επιτροπή Ένβη και θα της δώσω το λόγο. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, πέρσι η Κομισιόν παρουσίασε μια ανακοίνωση καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια ευοικονομία για την Ευρώπη και Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή, η Επιτροπή μας να εκδώσει μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Φυσικά η αρμόδια της Επιτροπή είναι Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ότι το, η αναζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κάτι που πρέπει όλοι να το υποστηρίζουμε και θέλουμε μια οικονομία που να βασίζεται πράγματι στις ανανεώσιμες πηγές, δεν τον φυσιτούμε αυτό, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι όταν κάνουμε αυτή την αλλαγή και από τα ρεκτά καύσιμα μεταβούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν μιλάμε για βιομάζα, θα έχουμε συγκρούσεις και ήδη έχουμε μια τέτοια κατάσταση σε σχέση με το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι της βιομάζας. Και επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και συγκρουόμενα συμφέροντα, κυρίως όταν πρόκειται για τη ζήτηση για δάση και για γη. Η αυξανόμενη ζήτηση για γη ήδη οδηγεί στην καταστροφή των δασών και της βιοπικιλότητας και Υπάρχουν και συγκρούσεις για την κατάκτηση των χειών. Έτσι λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδοτησή μου εστιάζομαι ιδιαίτερα στο εξή ότι χρειαζόμαστε ένα ορθό πολιτικό πλαίσιο για να λάβουμε όλα αυτά τα θέματα υπόψη. Όχι μόνο οικονομικής βιωσιμότητας, δηλαδή βιοοικονομία για την Ευρώπη, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε και στους παράγοντες της κοινωνικής ε, και οικολογικής αηφορίας. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα λοιπόν είναι ότι ε, το ποσό της ε, βιώσιμης βιομάζας από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιθανότητα ποτέ δεν θα αρκέσει για να καλύψουμε τη σημερινή ζήτηση σε ενέργεια και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές και πιθανότατα σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι η εξάρτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τι αγωγέ θα αυξήσει την πίεση στι παγκόσμιε συμφωνίε, όπω είναι η Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, το RED, και ότι η ε, ευξενόμενη ζήτηση προϊόντων ξυλία θα μπορούσε να προωθήσει παράνομη υλοτοπία και να επιδυναμώσει τι εθελοντικέ συμφωνίε εταιρική σχέση υπό του FLEGT. Κάτι που θα ήταν ε, καταστροφικό. Επίσης, ανησυχούμε για την, παράγοντε παράγοντες έμεσης αλλαγής χρήσης της γης, για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, το iLook. Και υπάρχει ανάγκη η Κομισιόν να προτείνει μια οδηγία πλαίσιο για τη βιομάζα που να καλύπτει όλες τις εφαρμογές της βιομάζας ενέργεια, καύσιμα, υλικά, χημικά και να εισαγάγει μια ιεράρχηση των ειδών βιομάζας. Με μια τέτοια ιεράρχηση, μια τέτοια ιεραρχία θα σημαίνει βασικά ότι δεν θα πρέπει να καίμε πράγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο, είτε για τροφή, για κατασκευές ή για άλλους σκοπούς ε, πέρα από το να πάρουμε την ενέργεια από τα ξύλα, το χάρη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολλαπλές χρήσεις, αλλά θα πρέπει να ξεκινούμε με την πιο πολύτιμη χρήση της βιομάζας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο επίσης και βέβαια η ζήτηση για τη βιομάζα στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα αυξήσει και την επιστηστική ανασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γνωρίζουμε την έννοια του land grabbing, της διαρπαγής της γης, αλλά Επίσης, ε, ήδη υπάρχει επίπτωση και στις τιμές των τροφίμων και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει τη σύσταση του δικού συγητή για το δικαίωμα στην τροφή για την ε, διασφάλιση της επιστικής ασφάλειας. Και επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί και η κλιματική αλλαγή. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι χρειαζόμαστε διεθνή πρότυπα νομικώς δεσμευτικά για όλους τους το, τομείς χρήσεων της βιομάζας ε, καθώς και κριτήρια ε, διαχείρισης, βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνάψει πολυμερείς συμφωνίες, κυρίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και συναφιδεσμική και τεχνική συστήριξη για να εξασφαλίσει τις βιώσιμες χρήσεις της βιομάζας. Αυτά είναι τα σημεία που περιλαμβάνονται στο πολύ περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων ε, για αυτή τη γνωμοδότηση. Στη... Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, το χάρη, δατοκαλλιέργεια, χρήση του νερού και των ε, παρακτονιδάτων και ξέρουμε ότι πολλά έλλη καταστρέφονται για να δημιουργηθούν ε, για γερατοκαλλιέργειες ε, και επίσης ε, ο πυθμένας της θάλασσας καταστρέφεται κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα και αυτά είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη γνωμοδότηση και Πιστεύω ότι όλη η έννοια των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Ε, έχουμε πολύ περιορισμένη εικόνα εδώ για τη βιομάζα στην ανακήρυξη της Κομισιόν. Δηλαδή κάνει λόγο μόνο για την οικονομική χρήση της άμεσης εκμετάλλευσης της βιομάζας, αλλά υπάρχουν και πολλές ε, αξίες ε, στα... αν αφήσουμε τα οικοσυστήματα και τα δάση ως έχουν και τα ψάρια στη θάλασσα, στο νερό αν θέλετε. Και φυσικά έτσι θα έχουμε καθαρό αέρα να αναπνεύσουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προσθέσουμε και αυτά τα στοιχεία στην γνωμοδότηση. Θα ήθελα βέβαια να ακούσω και τους συναδέλφους αν ε, έχουν κάποιες σκέψεις για το θέμα αυτό, αν θέλουν να καταθέσουν κάποιες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο. Merci ε, beaucoup. Oui, Monsieur Neusser, vous avez la parole. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Λέβιν για την έκθεσή της είναι πάρα πολύ καλή έκθεση εμείς δεν θα υποβάλουμε καμία τροπολογία το λέω ήδη από τώρα εκείνο το οποίο επίσης θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στη βιωσιμότητα όλων των μέτρων. Πώς ορίζεται η βιωσιμότητα. Η οικονομία, οικολογία και, κοινωνική παρά, παρά, και κοινωνικές παράμετροι, όλοι αυτοί οι παράμετροι, παράγοντες πρέπει να εναρμονίζονται. Στα, στις παραγράφους λοιπόν 4, 5 και 6 λέγεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε προβλήματα με μεγαλύτερη βιομάζα στις αναπτυσσόμενες χώρες και με την ε, αρπαγή ούτε με την αρπαγή της γης ότι θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί να μην βάλουμε σε δύσκολη θέση τους λαούς των αναπτυσσομένων χωρών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και το λέει βέβαια η έκθεση. Ίσως θα μπορούσε να γίνει πιο ισχυρή έντονη διατύπωση στα σημεία αυτά. Είναι και πολύ καλό που λαμβάνεται υπόψη η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών εδώ. Τώρα για την παράγραφο 6 πιο ειδικά ε, ε, μας αρέσει ιδιαίτερα ίσως είναι φιλόδοξοι στόχοι που αναφέρονται εδώ αλλά σε τελευταία ανάλυση γιατί να μην είμαστε φιλόδοξοι αυτή είναι η δουλειά μας ως Επιτροπής χαιρετίζουμε την έκθεση Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ ο λόγος στην Κομισιόν ο κ. Πολ και ο Ντομ Ντότ εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κ. Πορπρεσέ. Είναι και ο κ. Τόμ Ντότ, ο κ. Πρεσέ. Ελπίζω να μην <laughs> σας στενοχωρώ πολύ. Η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου στην στρατηγική για την ε, βιοοικονομία καθώς και τις ε, προσπαθίες σας να διατυπώσετε θέση επί του θέματος. Συμφωνούμε με την κεντρική ιδέα σας, δηλαδή με το ότι η βιοοικονομία πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα επί ποικιλίας θεμάτων. Οι τρεις αυτοί παράγοντες απαιτούν ακριβώς τη διατύπωση μιας συνολικής προσέγγισης στην οποία θα συνενέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πρέπει επίση να βελτιώσουμε την κατανόηση του προβλήματο από την κοινωνία μα γενικότερα και τι βασικέ έννοιε τη βιοοικονομία. Το λέω αυτό διότι είναι επιτροπή για την βιοοικονομία που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει και θέματα διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εννοείται ότι θα προσληθεί ως παρατηρητής στην Επιτροπή Βιοοικονομίας ε, μαζί βεβαίως και με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύσκεψη θα λάβει χώρα φέτος τον Ιούνιο. Καλό θα ήταν παρόμοιες επιτροπές να δημιουργηθούν και σε κρατικό, σε εθνικό και σε υποκρατικό επίπεδο. Συμφωνώ ότι χρειάζεται επαγρύπνηση για την παρανομή υλοτομία, το δικαίωμα στον επιστησμό, τον σεβασμό για τρέχουσες ε, συνθήκες όπως η CBD, η FLECT και εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της βιοοικονομίας με τρόπο που θα έχει θετικές επιπτώσεις εν προκειμένου αλλά και σε άλλους τομείς. Πολλά συναφή ζητήματα ήδη συζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας, στην εφαρμογή του προγράμματος έρευνας στο πλαίσιο του Οριζοντα 2020. Πρόκειται για έρευνα η οποία θα διαβατήσει κρίσιμο ρόλο στη διατύπωση της μελλοντική μας πολιτική. Διατύπωση την οποία φυσικά θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο με την έκθεσή του. Όσον αφορά τώρα την εισαγωγή βιομάζας, να τονίσω ότι χρειαζόμαστε πολιτικές αποτερικής χρήσης της βιομάζας. Έτσι θα έχει νόημα η προσπάθεια για να μειώσουμε τις πιέσεις στο περιβάλλον και στην βιοποικιλότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, δύο λόγια για τα δεσμευτικά πρότυπα αηφορίας στον τομέα της βιομάζας. Η Σχετική Επιτροπή καταρτίζει αυτά τα πρότυπα σε συνεργασία με τον Άιζο και στο πλαίσιο της βιώσιμης επιστημικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα. Πιστεύω ότι έτσι θα έχουμε κάποια μέτρα αναφοράς στο μέλλον. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Ξαναδίνω τον λόγο στην κυρία για να συνοψίσει. Ευχαριστώ. ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και ευχαριστώ και στην Κομισιόν για τα σχόλιά σας επί του σχεδίου νομοδότησης. Όλα αυτά ενισχύουν την εντύπωσή μου ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Ευελπιστώ ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί. Με πρόθυμη να συζητήσω με όποιον συνάδελφο το επιθυμεί και εκτός αυτής της συνεδρίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε λοιπόν την λήξη αυτής της συνεδρίασης. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Συνεχίζουμε πλέον και κλεισμένων των θυρών μεταξύ συντονιστών. Κατά τη διάρκεια αυτή τη συνεδρίαση, οι μόνοι που μπορούν να είναι παρόντε είναι οι βουλευτέ, οι βοηθοί του, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και οι υπάλληλοι τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ λοιπόν όλου του άλλου που δεν ανήκουν σε κατηγορίε να αποχωρήσουν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να συνεχίσουν και αυτή τη συζήτηση του εκτό αιθούση. Η συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα συνεχιστεί αύριο 9 ώρα το πρωί, στην ίδια αίθουσα. Με την ε, μεικτή συνεδρίαση Επιτροπών Εθνικών Κοινοβουλίων όσον αφορά την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη και τον συντονισμό των δωρητών.